Και περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης της απόψινής μας συνεδρίασης που είναι η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αδιέξοδο σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού υπαριθμών 1049 κάθετος 2001. Και θα δώσω τον λόγο στον Επίτροπο Μπορτ και πάλι. Παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω την ακόλουθη δήλωση. Στις 30 Απριλίου 2008 η Κομισιόν υπέβαλε μια πρόταση για μια αναδιατύπωση της του κανονισμού 1049-2001. Εφόσον εκκρεμούσε η πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την θέση σε ισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας υπέβαλε στις 21 Μαρτίου 2011 η Κομισιόν μια δεύτερη πρόταση ε, χωριστή αλλά συμπληρωματική στην πρώτη. Στόχος ήταν ε, να συμφωνεί, να συνάδει με τη νέα συνθήκη ο κανονισμός και με τον Ευρωπαϊκό ε, Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εφόσον η συνθήκη είναι δεσμευτική για τα θεσμικά όργανα όταν προτείνουν νόμους και για τα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν νόμους. Η πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 15 ε, Δεκεμβρίου 2011 περιλαμβάνει πολλές ε, τροπολογίες για διάφορα τμήματα του κανονισμού που η Κομισιό ε, δεν πρότεινε την τροποποίησή τους. Κατά την άποψη της Κομισιόν, οι τροπολογίες αυτές δεν είναι συμβατές με τις διοργανικές συμφωνίες του παρελθόντος η Κομισιό ανέφερε τη θέση της σε σχέση με τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανακοίνωση ε, για τα μέτρα που λήφθηκαν σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου ε, στο Δεκέμβριο ε, στην Ολομέλεια του 2011. Σύμφωνα με την τακτική νομοθετική διαδικασία η πρόταση της Κομισιόν και η θέση πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζονται από το Συμβούλιο. Το επόμενο βήμα σε αυτή τη διαδικασία είναι η οθέτηση μιας κοινής θέσης από το Συμβούλιο. Η Δανική Προεδρία προσπάθησε να επιτύχει μια συμφωνία σε έγκαιρη δεύτερη ανάγνωση. Η Κομισιό υποστήριξε τις προσπάθειες της Προεδρίας, αλλά κατά την άποψη της Κομισιό ανεπαρκής ο χρόνος αφιερώθηκε ε, στον ε, τριμερή διάλογο και στη συζήτηση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Αυτό το αποτέλεσμα λόγω έλλειψης ε, επαρκούς χρόνους για συζήτηση ε, δεν μπόρεσε ε, να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα εφικτό. Είμαστε ανοιχτοί για μια συζήτηση με όλους τους ε, κλάδους των νομιθετικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιό όμως επιμένει πάνω στην ανάγκη να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη κατάλληλης προστασίας άλλων νομοθετικών εγγράφων. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη προστασίας άλλων σημαντικών δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων και να δούμε ποια είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία θα μπορούσαν να φυγούν. Σας ευχαριστούμε για αυτή την δήλωση τοποθέτηση εξ ονόματος των ομάδων. Η κυρία Ρενάτε Ζόμερ είναι η πρώτη που θα παρέμβει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η αναθεώρηση του κανονισμού 1049 κάθετος 2001 για την πρόσβαση του κοινού των πολιτών σε έγγραφα τώρα έγινε μια τέλειωτη ιστορία πραγματικά γιατί δεν προχωρεί αυτό το χαρτοφυλάκιο και δεν προάγεται. Όχι επειδή από πλευράς του εισηγητή δεν υπάρχει η πρόθεση να υπάρξει κάποια πρόοδος. Επειδή επιμένει σε κάποιες συμβιβαστικές ε, ε, λύσεις και γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχουν εδώ παραβιάσεις νομοθεσίας και φυσικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν είναι κάτι τέτοιο αποδεκτό ακόμα και οι περίεργες ε, απόψεις ε, για δημοσιοποίηση οποιονδήποτε στοιχείων από οποιαδήποτε θεσμικά όργανα είναι ακριβώς το αντίθετο εκείνου του που συμβαίνει σε σχέση με τον ευκταίο στόχο που θέλουμε εμείς να επιτύχουμε διότι πραγματικά τα σημαντικά έγγραφα είναι εκείνα τα οποία δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Αν τις θεμελιώδεις πληροφορίες ε, δεν τις δημοσιεύουμε, τότε οι πολίτες μας ε, δεν θα έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και στα θεσμικά της όργανα και ούτε θα την κατανοούν εκείνη και τα θεσμικά όργανα. Κάτι τέτοιο θέλουμε. Ταυτόχρονα και το έργο μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθίσταται αδύνατο πλέον. Αν σε κάθε συζήτηση που γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να δημοσιεύσουμε τα πάντα και να πρωτοκολούνται τα πάντα, τότε αυτό θα ήταν προ όφελο του Κοινοβουλίου. Φυσικά όχι. Είναι αυτό προ όφελο των πολιτών μα λοιπόν ω κατάσταση. Όχι. Η δική μου ομάδα πάντα ήταν υπέρ του ότι οι μηχανισμοί και η νομοθεσία στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να είναι διαφανέστεροι και πιο ε, αποτελεσματικοί. Φυσικά θέλουμε να έχουν πρόσβαση οι πολίτε σε έγγραφα. Όμω γνωρίζουμε από την άλλη πλευρά επίση ότι αυτή η πρόσβαση πρέπει να αριθμίζεται με μια ε, συνετή ισορροπία Αφενός σε σχέση με την προστασία των δεδομένων που πρέπει να διασφαλίζεται, αφετέρου για εκείνα τα θέματα όπου είναι αναγκαίο να υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα δημοσιοποιούνται. Και αυτό θα πρέπει να εξεύρει ισορροπία προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων. Και σε δυσχερείς συζητήσεις και με το Συμβούλιο και την Επιτροπή καταστήσαμε σαφή αυτή την στοχοθέτηση. Από πλευράς όμως εισηγητού δεν λαμβάνεται αυτό υπόψη. Και αγνοεί το στόχος της μεγαλύτερης διαφάνειας και της προστασίας των πολιτών επιλέγονται σημεία τα οποία δεν μπορούν να είναι αντικείμενο ε, μιας τέτοιας ρύθμιση, γιατί τη δημοσιοποίηση ε, στοιχείων ε, εκκρεμουσών υποθέσεων για παράδειγμα όπως και στους τριμερεί διαλόγους που επιβαρύνουν, επιβαρύνονται με αυτά τα θέματα. Έτσι ωστόσο η διαδικασία επίτευξης του στόχου είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί. Ακόμα και η άσκηση λομπιστικής δραστηριότητας είναι κάτι το οποίο δεν δεν μπορούμε να δεχτούμε Επίσης η προστασία της ε, πνευματικής ε, ε, ιδιοκτησίας. Επίσης σε σχέση με θέματα δημοσιοποίησης όσον αφορά προσωπικά θέματα. Όμως δεν πρέπει να δώσουμε την ιδιωτική ζωή, την, τα στοιχεία του ιδιωτικού βίου των πολιτών σε ισοπεδωτική δημοσιοποίηση. Καθώς επίσης και τα θέματα τα οποία πρέπει να δημιουργήσουν πρόσθετη αξία για τους πολίτες μας και να δεχθούμε λοιπόν μέσω αυτή τη προσπάθεια την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ ο εισηγητή να το δεχτεί αυτό. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Έχει τον λόγο εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω ότι και η θέση της κυρίας Ζόμερ ε, αντιπροσωπεύει και τη θέση ε, του εισηγητού αλλά και τη θέση του, της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου. αυτή η αναθεώρηση του κανονισμού δεν είναι ικανοποιητική όπως είπε και η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πρέπει να πω ότι οι προσπάθειες της Προεδρίας και οι δικές μας δυναμητίστηκαν πλήρως από την παρασκηνιακή εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ε, πραγματικά δεν βοήθησε καθόλου την εργασία ε, του Κοινοβουλίου. Ο αρμόδιος Επίτροπος δεν εμφανίστηκε καν ενώπιον της Επιτροπής Λίμπε που τον είχε καλέσει. Όλες οι προτάσεις συμβιβαστικών λύσεων, όλες οι τροπολογίες ε, που συζητήθηκαν στον τριμερή διάλογο, δεν, από αυτές καμία δεν έγινε δεκτή. Κοιτάξτε, εγώ είμαι έτοιμος να δημοσιοποιήσω ε, τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και είμαι βέβαιος ότι και η Ιδανική Προεδρία θα μπορούσε να κάνει το ίδιο. Ε, και νομίζω ότι πρέπει να δημοσιευθούν τα έγγραφα αυτά έτσι ώστε να αποφασίσει επιτέλους να κάνει και τη δουλειά του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για τους ε, πολίτες. Η συνθήκη της Ευρώπης, έχει, συγγνώμη, η συνθήκη της Λισαβόνας έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες όσον αφορά την πρόταση του κοινού στα έγγραφα και ο Γενικός Εισαγγελέας πολύ σωστά ανέφερε ότι σε μία δημοκρατική κοινωνία η σωστή λειτουργία μπορεί να γίνεται μέσα από σωστές διαδικασίες. Έχουμε λοιπόν τον Γενικό Εισαγγελέα ο οποίος ε, μαζί με το Κοινοβούλιο προσυπογράφει τη θέση ε, για μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίσης ε, θα πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής σε, σε όλα τα θεσμικά όργανα και λοιπά όργανα και υπηρεσίες. Χρειαζόμαστε νομοθετική διαφάνεια Χωρί χωρίς καμία ε, ε, εξαίρεση κατά τα λοιπά βεβαίως το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ξανακαθίσει το τραπέζι διαπραγματεύσεων και να βρει συμβιβαστική λύση παρά τις ε, προσπάθειες και της κυρίας Ζόμερ και του υποφαινόμενου δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Ας προχωρήσουμε όμως, ας δουλέψουμε όλοι μαζί. Όμω, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να δουλέψει μόνο του, χρειάζεται και την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Εάν παραμείνει αυτό το αδιέξοδο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πολλοί θα είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι πολίτε οι οποίοι θα απεμπλακούν εντελώ από την Ευρωπαϊκή διαδικασία. Το Κοινοβούλιο όμως δεν είναι ε, δυνατόν να είναι συνένοχο σε μια τέτοια άσχημη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάσμα. Ζήτησε τον λόγο τώρα η κυρία Σαρτζεντίνη, παρακαλώ. Ehm, Ευχαριστώ πολύ. Λίγο πιο πριν αναφερθήκαμε κύριε Πρόεδρε ε, στο πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης και τη θέση ψυχόλου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Και μιλήσαμε και για τον τρόπο με τον οποίο ε, οι πολίτες βλέπουν, αντιλαμβάνονται την Ευρώπη. Ορίστε, εδώ έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε τον σκιώδη συγητή του ΕΛΚ που μας λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει το απόρριτο ή εμπιστευτικότητα ε, και κάποια έγγραφα να γίνονται δημόσια. Όμως ε, μονάχα κάποια έγγραφα τα οποία αφορούν δημόσια υγεία ή ε, που μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλη αναστάτωση στη κοινωνία θα πρέπει να παραμένουν κάπως μυστικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε αυτήν την ε, κρυψίνια διότι συμφωνώ με τον εισηγητή τότε θα δημιουργήσουμε μεγάλη δυσπιστία στον κόσμο. Ε, θα πρέπει από κοινού να δράσουν το Συμβούλιο και το ε, Κοινοβούλιο και θα πρέπει να έχει το κοινό ελεύθερη πρόσβαση στα έγγραφά μας, να ξέρει τι κάνουμε και γιατί συζητάμε. Υπάρχουν χώρες όπως η Δανία ή όπως η χώρα η δικιά μου, οι κάτω χώρες, ε, οι οποίες έχουν τέτοια παράδοση και θα μπορούσε να ακολουθήσει το, η Κομισιόνα το παράδειγμα των χωρών αυτών στο κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο επανειλημμένα επιμένει προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά φαίνεται ότι ε, δεν ε, έχετε αρκετή εμπιστοσύνη στους πολίτες μας. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιώργος Παπα-Νικολάου παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για την εφαρμογή του προγράμματος Στοχόλμης αναφερθήκαμε στο ζήτημα της αναθεώρησης του κανονισμού για την πρόσβαση στα έγγραφα και όλοι συμφωνήσαμε ότι έχουμε μείνει πίσω στο θέμα αυτό και πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι πράγματι δημοκρατική υποχρέωση και πηγάζει από τη συνθήκη της Λισαβόνας, υπόθηκε ήδη, η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και είναι ζήτημα λογοδοσίας να συμβαίνει αυτό, κανείς δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος πολύ δε περισσότερο εις βάρος του δημόσιου βίου και των προσωπικών δεδομένων. ο επίτροπος σήμερα ο επίτροπος borg τοποθετήθηκε σωστά. τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να μπαίνουν, ούτε να μπαίνουν σε ζυγαριά ούτε να αποδεχόμαστε τη θυσία κάποιων από αυτά προς όφελος κάποιων άλλων. με δύο λόγια αντισταθμίζεται πλήρως η προσβολή του δημόσιου συμφέροντος από την ανάγκη πλήρης δημοσιοποίησης όλων των εγγράφων. αντισταθμίζεται η έκθεση στη δημοσιότητα στοιχείων πολιτών πολλό δε μάλλον ανηλίκων για λόγους διαφάνειας προφανώς η διατήρηση αυτής της ισορροπίας δεν είναι πάντα εύκολη αυτό το γνωρίζει και ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές δεν ήταν καθόλου εύκολη η πορεία μέχρι εδώ πολλές ήταν οι διαφωνίες πολλές ήταν οι προστριβές αυτό καταμαρτυρούν άλλωστε και τα πέντε χρόνια από την αρχική ανακοίνωση της επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού παρακολουθώντας ωστόσο την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων διαπιστώνεται και μια σχετική έλλειψη των προβλέψεων καταγραφής στο μητρό των ευαίσθητων εγγράφων και θα ήθελα με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης και με την παρουσία του επιτρόπου να ρωτήσω και να έχω μια απάντηση αν αυτό είναι δυνατό για ποιο λόγο κύριε επίτροπε για ορισμένα έγγραφα δεν είναι καν καταγεγραμμένα στο σχετικό μητρό άσχετα αν παρέχεται ή όχι η πρόσβαση σε αυτά. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. επόμενο αγορητή ο κύριο Κλοντ Μωράη Thank you, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να, να στηρίξω απολύτως τον εισηγητή μας, τον κύριο Κάσπαν, και να συμμεριστώ την ε, απογοήτευσή του για την έκβαση ε, της ε, συζήτησης. Καλό είναι που ξανασυζητάμε σήμερα για να δούμε αν μπορέσουμε, αν έχουμε ρεαλιστικά πιθανότητες να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε ε, αυτό το ζήτημα. Ε, πρέπει να έχουν πρόσβαση οι πολίτες μας ε, στα έγγραφα. Έχουμε άλλωστε και την πρώτη συμφωνία της 12ης ε, του, του ε, Δεκεμβρίου του 2011. Ε, τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι πιστεύουμε στη λογοδοσία και ότι πιστεύουμε και στην πλήρη διαφάνεια. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνουμε μεγάλη δυσπιστία και βεβαίως θα συνεχιστεί η δυσπιστία και η αυξανόμενη απογοήτευση των πολιτών όταν ε, δουν ότι δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά ε, και την ε, διαφάνεια. Το 2008 ήδη είχε ξεκινήσει η συζήτηση και βεβαίω τότε είχαν συζητηθεί κάποιες πληροφορίες οι οποίες πρέπει να είναι μυστικές γιατί παρουσιάζουν μεγάλο, μεγάλη σημασία για το κοινό συμφέρον. Κατά τα άλλα όμως δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να δυναμητιστεί αυτή ε, η δημοκρατική διαδικασία. Ο συνάδελφος Μάικλ Κάσμαν έχει δίκιο όταν λέει ότι οι πολίτες πρέπει να ξέρουν τι γίνεται στο σώμα εδώ, ε, μια και είναι, ε, δρούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βουλευτές εκλεγμένοι εξ ονόματος των πολιτών και εκλεγμένοι με την ψήφο των πολιτών που μιλούν εξ τους και επομένως δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουν τι γίνεται εδώ μέσα. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει κανείς ε, να καταλάβει και τι γίνεται στο μυαλό της Κομισιόν και του Συμβουλίου και που δεν καταλαβαίνουν ένα τόσο απλό και προφανές πράγμα. Σας ευχαριστούμε συνάδελφος κυρία Ιντφέλτ παρακαλώ. Ε, yes, thank you, Chair. Um, I would like to... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Σόμερ που ήταν πραγματικά η προσωποποίηση του Σερ Χάμφρι σε σχέση με αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι άκουσα κάποιον να λέει σε αυτό σε αυτή την ολομέλεια ότι δεν πρέπει να δίνονται υπερβολικές πληροφορίες στους πολίτες διότι αυτό θα δημιουργήσει σύγχυση σε αυτούς. Αυτό είναι κάτι από μια τηλεοπτική φάρσα. Δεν μπορεί να είναι πραγματικό κάτι τέτοιο. Να σας ακούμε με αυτόν τον τρόπο κυρία Σόμερ είναι απίστευτο. Και δεν είναι το ε, εγχείρημα διπλωματών όπου ε, επικρατεί η ας το πω έτσι απόκρυψη στοιχείων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί σε μια πολιτική ένωση για τους ε, πολίτες και οι πολίτες ζητούν και κραυγάζουν να υπάρξει διαφάνεια διότι η διαφάνεια είναι εκείνο το απαραίτητο στοιχείο για τη λογοδοσία που είναι απαραίτητο πάλι με τη σειρά του στοιχείο για μια ε, δημοκρατική τάξη πραγματών. Ακούμε να λέει πολλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο που θέλγονται από αυτά. Πολύ λόγο κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκατασταθεί, λέει, η εμπιστοσύνη των πολιτών. Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημαθεί στην Επιτροπή ότι συζητούμε στην Ολομέλεια εδώ από αυτού του θέματο Να αποφύγουν τι συζητήσει μεταξύ του. Κύριε Επίτροπε, συγγνώμη, κύριε Επίτροπε, συγγνώμη. Κύριε Επίτροπε, πραγματικό, πραγματικά σας παρακαλώ να φορέσετε τα ακουστικά σας και να προσέξετε την ομιλήτρια. Θα έπρεπε να προσέχουν αυτά τα οποία λέγονται στην Ολομέλεια. Εμείς Ακούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει συχνά να αποκατασταθεί λέει η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όμως δεν υπάρχει πολιτισμός διαφάνειας, κουλτούρα διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς είναι δυνατόν να ε, υπάρχουν προσφυγές στα δικαστήρια όταν αρνείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την δημοσιοποίηση στοιχείων και θα πρέπει να γίνουν ε, τέτοιου είδους προσφυγές στα δικαστήρια. Όμως το άκτα το έχετε ακούσει ως συμφωνία. Αν θέλετε μια απόδειξη του τι γίνεται όταν υπονομεύονται τα σχέδιά μας ε, για διαφάνεια, η υπόθεση άκτα είναι ιδανική περίπτωση. Θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει διαφάνεια και αποκαλύπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο είναι το δυνατόν λιγότερα στοιχεία. Παρακαλώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας για να αποτροχοπεδηθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο. Σας ευχαριστούμε κυρία Όκεν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου οι πολίτες δείχνουν αυξανόμενη δυσπιστία προς εμάς αλλά και γενικότερα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερως δε ε, δείχνουν δυσπιστία προς την Κομισιόν η οποία όμως φαίνεται να αγνοεί αυτό το ε, στοιχείο και να αγνοεί επίσης ε, ότι να αγνοεί το γεγονός ότι και η Κομισιόν βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών. Ο πολίτης πρέπει να είναι το επίκεντρο των διαδικασιών μας. Ε, και άλλωστε μην λησμονούμε τη συνθήκη της Λισαβόνας μέσα από την οποία ε, διαβεβαιώσαμε τους πολίτες ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Εγώ θυμάμαι τη Δανική Προεδρία και πολύ καλά μάλιστα και ε, μου είπαν ότι τους είχαν πει, ε, στη Δανική Προεδρία δηλαδή, ότι τους είχε πει η Κομισιόν ότι δεν είναι και πολύ καλή ιδέα να κινήσουν πολύ το ε, ζήτημα. Όμως έχουμε ε, και μία ε, τάση γενικώ ε, να ε, αφήνουμε αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα πίσω μας ή να τα κρύβουμε. Μα πηγαίνουμε προς μια νέα εποχή κύριε Επίτροπε και επομένως δεν έχει καμία έννοια ε, να προσπαθούμε να έχουμε στην Κομισιόν ας πούμε μηδενικό επίπεδο λάθους ε, εάν ε, δεν υπάρχει μια δημοκρατική συζήτηση ή δημοκρατικές διαδικασίες όλοι κάνουμε λάθη και είναι καλύτερα να έχουμε διαφάνεια παρά να προσπαθούμε μονάχα να φτάσουμε στο μηδενικό επίπεδο λάθους. Μας είχατε υποσχεθεί και ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών, ακόμα το περιμένουμε. Σα ευχαριστούμε κυρία Κοράτσα Μπιλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα είναι απαραίτητη για να υπάρχουμε άνοιγμα και να συμμετέχουν οι πολέτες στην νομοθετική διαδικασία. Ήρθε η ώρα ε, να λήξει αυτό το αδιέξοδο. Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο και καλό την Κομισιό το Συμβούλιο και την Προεδρία να κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι και να αρχίσουν ε, τις διαπραγματεύσεις με επικοδομητικό πνεύμα. Ο νέος κανονισμός θα πρέπει στο τέλος της θητείας να υιοθετηθεί. Όχι, όχι, δεν θέλουμε συμβιβασμούς πάση θυσία, αλλά να ενισχύσουμε την διαφάνεια με υπεύθυνο και σαφή τρόπο την, ε, εφόσον η Βρυξέλλες είναι μακριά από το σπίτι μας, πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, ε, τα όργανα για να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη στους ε, θεσμούς. Τι, να έχουμε διαφάνεια με μυστικότητα, τι φοβόμαστε, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις και το θέμα είναι περίπλοκο. Η προστασία των δεδομένων, η ακαιρεότητα ε, θα πρέπει ε, να τηρούνται. Αλλά, αγαπητή Σοφή, η δημόσια πρόσβαση δεν σημαίνει Wikileaks θα εξακολουθήσω και εγώ να δεσμεύομαι για την διαφάνεια, την υπευθυνότητα, να δημοσιεύω τους λόμπιστ που συναντώ το πρόγραμμά μου και να αποφεύγω την μυστικότητα. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ξέρουν πώς λαμβάνουμε αποφάσεις στο όνομά τους που επηρεάζουν τις ζωές τους. Ανοίξουμε τις πόρτες μας και ας τους επιτρέψουμε όχι μόνο να παρακολουθούν αλλά και να συμμετέχουν, ότι είναι μέρος μιας κοινότητας όπου λαμβάνονται αποφάσεις δημοκρατικά. Να τους δείξουμε ότι πραγματικά αντιπροσωπεύονται. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και σιωθετήσουμε αυτό τον κανονισμό. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ, δέχεστε μια ερώτηση από την κυρία Ιντφελτ. Παρακαλώ. Yes, thank you. Ε, Ευχαριστώ για να αρθεί μια παρανόηση. Δεν είπα ότι τα Wikileaks θα πρέπει αντί της ε, διαφάνειας ε, στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει να λειτουργήσουν, αλλά να είναι εκείνοι οι πολίτες ε, που θα λαμβάνουν υπόψη. Επίσης αυτά τα οποία είπατε θα ήθελα να πω ότι αντιφάσκουν σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν από την κυρία Σόμερ πιο πριν. Και θα ήταν πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε ποια θα είναι η θέση του ΕΛΚ στο τέλος. Ελπίζω ότι θα είναι η δική σας θέση η θέση του ΕΛΚ τελικά. Κυρία μπορείτε να απαντήσετε, παρακαλώ. I, uh, Απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Σόφη ε, που αποσαφήνισε το θέμα αυτό για το ε, Wikileaks γιατί ε, η χρήση συκοφαντικών δυσφημίσεων και τέτοιων μέσων δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Όσον αφορά το ΕΛΚ, θέλουμε μεγάλη διαφάνεια και μεγαλύτερο άνοιγμα και θέλουμε να ε, κλείσουμε αυτό το δημοκρατικό κενό με, το, ε, με τους πολίτες. Αλλά βεβαίως πρέπει κανείς να δει πολύ προσεκτικά τι γίνεται με την νομική βάση, τι γίνεται ε, όταν ας πούμε μιλάμε στους διαδρόμους μεταξύ μας ή όταν δίνουμε ο ένας ένα χαρτί με μια παρατήρηση στον άλλον και επίσης δεν χρειάζεται να μπούμε σε οποιαδήποτε, σε οποιοδήποτε ανταγωνισμό με την Κομισιόν. Θα πρέπει να εργαστούμε έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Η κυρία Βίκστρομ τώρα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή ουσιαστικά δεν ανήκει ως θέμα σε μια ανοιχτή σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα το 2013. Ουσιαστικά θα έπρεπε να είχε διεξαχθεί πριν από πολλές δεκαετίες. Το πρώτο ερώτημα το οποίο θα έπρεπε να διατυπώσουμε είναι ποιος είναι ο κάτοχος, ποιος έχει την κυριότητα αυτών των στοιχείων δεδομένων πληροφοριών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι. Οι ιδιοκτήτες που έχουν την κυριότητα είναι οι πολίτες και φυσικά έχουν το δικαίωμα να έχουν στη διάθεσή αυτά τα στοιχεία. Και δεν μπορεί να καθορίζουμε εμείς το τι θα γίνεται και μάλιστα με αντίθετο τρόπο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει με σαφέστερο τρόπο τον ρόλο προπομπού. Η απόκρυψη και η μυστικότητα δεν είναι το μέλλον και στη συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρεται ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λειτουργούν με το μεγαλύτερο ανοιχτό και διαφανέστερο πλαίσιο. Λυπούμε ότι είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαφορετική και σε σχέση με τα όσα έχουν γίνει και όλα αυτά δεν συνάδουν με μια πιο ανοιχτή, διάφανη Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ των πολιτών την οποία επιθυμούμε και στην οποία ελπίζουμε. Πρόεδρος, τώρα έχουμε την περίοδο συζήτησης με το Catch the Eye. Έχουμε και πάλι παρέμβαση της κυρίας Μπασέσκου. Παρακαλώ κυρία Μπασέσκου. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η πρόσβαση στα έγγραφα και δεδομένα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αποτελεί μια σημαντική εναλλακτική δυνατότητα για τους πολίτες να μπορούν οι πολίτες να ελέγχουν τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια μεγαλύτερη διαφάνεια θα ενδυνάμωνε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτά τα θεσμικά όργανα και θα διευκόλυνε τους πολίτες να καταλαβαίνουν καλύτερα πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις από αυτά τα θεσμικά όργανα. Θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση με μια ρύθμιση που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές πραγματικές ανάγκες ε, της πραγματικής ζωής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει ήδη την άποψή του σε σχέση με αυτή τη ρύθμιση. Όμως αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο και δεν προχωρούν τα πράγματα. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα και δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε μια προθεσμία 15 ημερών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι πολίτες μετά από ετοιμά σε τέτοιου είδου στοιχεία και έγγραφα. Ταυτόχρονα ταυτόχρονα όμως μια τέτοια προθεσμία θα πρέπει να καθορίζεται για να μπορούν όλα αυτά να λειτουργήσουν. Τώρα έχουμε και τις τελικές ε, δηλώσεις του Επιτρόπου Μπόργκ. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως θα αρχίσω λέγοντας σαφώς ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υπάρξει ε, ο φυστάμενος κανονισμός αναθεωρημένος. Πρόταση της Κομιζιό ε, είναι προς αυτή την κατεύθυνση να γίνει ο κανονισμός αυτός συμβατός με τη συνθήκη της Λισαβόνας και τον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι ε, για να έχουμε μια συμφωνία θα πρέπει οι δύο συνομοθέτες να διαπραγματευτούν και να συμφωνήσουν. Να υπενθυμίσω εδώ ότι ε, ε, δεν επέτυχε η ιδανική προεδρία να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό. Μια πλειονότητα κρατών μελών συμμερίζεται την άποψη της Κομισιόν και δεν υποστήριξε τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Η Κυπριακή ε, Προεδρία διερεύνησε την δυνατότητα να βρεθεί ένα κοινό έδαφος, αλλά συνεπέρανε ότι οι συνθήκες για ένα συμβιβασμό δεν επληρούνται. Και η τρέχουσα Ιρλανδική Προεδρία δεν πήρε περαιτέρω πρωτοβουλίες, αλλά αυτό είναι το παρελθόν. Θα πρέπει να ταινίσουμε το μέλλον και νομίζω ότι η Κομίσιο μπορεί να δεσμευτεί να ε, θέσει το θέμα με την επερχόμενη Λιθουανική Προεδρία, ούτως ώστε το Συμβούλιο να επανεξετάσει το θέμα και να, θα πρέπει τότε να οργανώσει διμερή ε, τρίλογο ε, για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Πρόεδρος, για διαδικαστικό, κύριος Κάσμαν παρακαλώ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό διαδικαστικό αυτό. Μια ναι, και το Ευρωκοινοβούλιο έχει απόλυτα αντίθετη άποψη σε σχέση με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις υπό την Δανέζικη Προεδρία και την Κυπριακή Προεδρία και είμαστε πρόθυμοι να ε, καταθέσουμε και να δημοσιοποιήσουμε τις δικές μας ε, τροπολογίες και προτάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει τις δικές της τροπολογίες και τις δικές της ε, προτάσεις σε σχέση με τη διατύπωση αυτή. Δεν έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Αν θέλουν όμως και ξαφνικά ο ε, εισηγητής δεν μπορεί να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, θα τα δημοσιοποιήσουν και ο λόγος είναι επειδή το, το Συμβούλιο πρέπει να έχει την πρώτη ανάγνωση που πρέπει να ολοκληρωθεί θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμφωνήσει μαζί λοιπόν, μα η να αποσυρει Επιτροπή. προτάσει. Δεν φοβουμε λοιπον οτι το προβλημα ειναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Δεν ήταν όμως για διαδικαστικό αυτή η ευρωπαικη επιτροπη ευχαριστω δεν ηταν όμω για διαδικαστικο αυτη η παρεμβαση Θα θεωρούσα ότι είναι μια ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η παρέμβασή σα. Κύριε Επίτροπε θέλετε να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση ή όχι. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι η έκκληση που κάνω είναι να, να προσβλέψουμε στο μέλλον και ότι η Κομισιόν θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό με την Λιθουανική Προεδρία. Η ήδη έχει αναφέρει την θέση της η Κομισιόν σε σχέση με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στην ανακοίνωση και σε σχέση ε, με τα όσα έκανε και αποφάσισε το Δεκέμβριο 2011 το Κοινοβούλιο. Ε, θα αναφέρουμε το θέμα αυτό στην Λιθουανική ε, Προεδρία και ελπίζω να υπάρξει μια επανεκκίνηση σε σχέση με το θέμα. Προεδρεύων, σας ευχαριστώ θερμά. Ολοκληρώνω τη συζήτηση εδώ. Η ψήφιση θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου τον Ιούνιο. Η επόμενη συνεδρίασή μας στην Ολομέλεια θα είναι αύριο Τετάρτη 22 Μαΐου στις 8.30 το πρωί. Πρώτο τμήμα μέχρι τις 14.00 και το δεύτερο τμήμα από 15.00 έως 22, 23.00. Έχει δημοσιευθεί η ημερησία διάταξη.